meine sehr geehrten damen und herren! Καθίστε κυρίε και κύριοι και κηρύσω την επανάληψη της συνόδου που διακόπησε στις 27 Μαΐου. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού ξεκινήσουμε τις εργασίες